Θα δούμε πόσο θα προχωρήσουμε στη συζήτηση και μετά θα δώσουμε συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την ε, εκλογή των κοσμητόρων. Χαιρετίζω τον ανεργία προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Πρωθυπουργό, κύριο Σαμαρά. Κύριε Σαμαρά, θα έχετε αμέσως τον λόγο. Παρακαλώ. κύριε πρόεδρε του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές θέλω κύριε πρόεδρε στην αρχή να σας συγχαρώ για την εκ νέου εκλογή σας αλλά και για τη συνέπεια την αγωνιστικότητα και τη δύναμη της πίστης σας στην ενωμένη ευρώπη. θέλω επίσης να συγχαρώ τον παρευρισκόμενο κύριο μπαρόζο για την προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό ιδεώδες και την τόσο πετυχημένη παρουσία του ως Προέδρου της Επιτροπής. Και οφείλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και το νέο τρόπο εκλογής πρότεινε στην Ευρωβουλή την υποψηφιότητα του Ζων Κλοντ Juncker ενός αφοσιωμένου Ευρωπαίου εγνωσμένης αξίας, πείρας και ικανότητας. Αγαπητοί φίλοι, είναι για μένα ιδιαίτερη συγκίνηση σήμερα να βρίσκομαι εδώ σε ένα χώρο γνώριμο που το νιώθω πραγματικά σαν να είναι το σπίτι μου. Υπήρξα Ευρωβουλευτής σε αυτά ακριβώς τα έδρανα που βρίσκεστε εσείς, ακριβώς πριν 10 χρόνια. Πάλεψα για τα ίδια ιδανικά, για το κοινό μέλλον δηλαδή των λαών της Ευρώπης και μάλιστα πολλά από αυτά που σήμερα θεωρούνται δεδομένα για όλους τότε ήταν αδιανόητα για οποιονδήποτε γιατί το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ζωντανό έχει ελλείψεις έχει αδυναμίες προχωράει άνεσα Άνεσα, αλλά προχωράει και μάλιστα πολλές φορές θα έλεγα με θεαματικά άλματα. Και αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει μόνον αν δει τα πράγματα από κάποια απόσταση. Πράγματι υπάρχει αλματώδης πρόοδος από τη μια δεκαετία στην άλλη μέσα σε μια γενιά έγιναν όσα λίγοι πίστευαν και ακόμα λιγότεροι περίμεναν μερικές δεκαετίες πριν. Και ο ρυθμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιταχύνεται συνεχώς. Με συγκίνηση λοιπόν σας καλωσορίζω όλους τους νέους συναδέλφους και εύχομαι καλή επιτυχία στην καινούργια σταδιοδρομία σας. Πολύ περισσότερο που σήμερα βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω τα αποτελέσματά μας της Προεδρίας μας, της Ελληνικής Προεδρίας. So Επιτρέψτε μου τώρα να, συνεχίσω στα αγγλικά. Οι προτεραιότητες μα για την εξάμεινη προεδρία μα ήταν οι εξή. Πρώτον, να αντιμετωπίσουμε τι ε, θεσμικέ ανεπάρκειε του ευρώ, όπω τις κατέδειξε η κρίση. Κυρίως να εμβαθύνουμε την Οικονομική Νομισματική Ένωση. Η επιτυχής κατάληξη του κανονισμού SRM για την ενιαία εξυγίανση, το μηχανισμό για την ενιαία εξυγίανση και η διακυβερνητική συμφωνία για το ενιαίο ταμείο εξυγίανση, SRF, αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προ την ολοκλήρωση τη Τραπεζικής Ένωση. Η νομισματική μα ένωση είναι τώρα πολύ καλύτερα εξοπλισμένη για να αποφύγει μελλοντικέ κρίσει και καλύτερα προετοιμασμένη για να τι αντιμετωπίσει εάν συμβούν. Τώρα για την απασχόληση και την ε, ανάπτυξη. Η έγκριση του νομοθετικού πακέτου για του ίδιου πόρου θα διασφαλίσει την έγκαιρη και σταθερή χρηματοδότηση των ενωσιακών πολιτικών. Η έγκριση νομοθεσία στα πλαίσια της ε, πράξης για την έννοια αγορά 1 και 2 συνέβαλε περαιτέρω στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Διευκολύνει και προασπίζει την οικονομική δραστηριότητα των πολιτών μας και των επιχειρήσεων. Να αναφέρω τα εξή. Πρώτον, τον κανονισμό για τις ε, ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο, την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση των δημοσίων προμηθειών, και την γνωστοποίηση μη χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Περαιτέρω, επετεύχθη σύμφωνια για τη συμμετοχή της Ένωσης στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Αυτό σημαίνει περισσότερη ρευστότητα για να αποκαταστήσουμε κανονική δανειοδότηση στην οικονομία, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες, που είναι το πιο σημαντικό τμήμα της οικονομίας μας. Σημαντικά θέματα επενδύσεων επίσης κατέληξαν επιτυχώς, ενώ σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υποδομών. Καλύτερη χρηματοδότηση, περισσότερη ευελιξία των αγορών, περισσότερη πρόσβαση στις αγορές για όλους, περισσότερη πρόσβαση στη ρευστότητα για τις μικρομεσαίες, περισσότερη διαφάνεια παντού στην Ένωση. Όλα αυτά είναι διαφορετικές πλευρές δύο βασικών αξώνων. Περισσότερη ενοποίηση και περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, καλύτερες προοπτικές για θέσεις εργασίας, απασχόληση, ανάπτυξη, ευημερία. Ιδιαίτερα σε περιόδους όταν η τεράστια ανεργία, τα τεράστια επίποδα ανεργίας απειλούν την έφραυστη κοινωνική συνοχή σε πολλά κράτη-μέλη. Τρίτον, διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόκληση, όχι μόνο για τον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά οπωσδήποτε για συνολικά την Ένωση με πολύ εκτεταμένες επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερα σημαντικά επιτεύγματα ήσαν πρώτον η αναθεώρηση του καταλόγου των χωρών που απαιτείται προξενική θεώρηση για να εισέλθουν οι πολίτες του στην Ένωση, επιτρέποντας έτσι σε πολίτες ε, περίπου 23 χωρών να ταξιδεύουν στην Ένωση χωρίς τραπεζική θεώρηση και δεύτερον η έγκριση της οδηγίας για τις συνθήκες ε, εισόδου και παραμονής πολιτών τρίτων χωρών στα πλαίσια των διαεπιχειρηματικών μεταθέσεων καθώς και ο νέος κανονισμός Frontex. Μεγάλη επιτυχία ήταν η έγκριση των στρατηγικών κατευθυντηρίων ε, μετά τη Στοκόνη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης που εστιάζει στην εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης στον τομέα του ασύλου, και τη διαχείριση των συνόρων και τη μετανάστευση. Και δεύτερον, η σύνδεση μεταξύ τη μετανάστευση και, ε, και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, δηλαδή συνεργασία με τρίτε χώρε, περισσότερα για περισσότερα κτλ. και η ανάπτυξη αποτελεσματική πολιτική επιστροφή, επανεισδοχή πολιτικών θεωρήσεων και συνεχής προσοχή στην προσπάθεια δημιουργία ενό αποτελεσματικού εσωτερικού πλαισίου ασφαλεία, Τέταρτον, η οριζόντια θεματική τη ελληνική Προεδρίας ήταν ο επανακαθορισμός και η επανεκκίνηση της ενωσιακής πολιτικής για τη θάλασσα από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένες της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ενέργειας. Βασικό στατικό στοιχείο είναι η στρατηγική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια της θάλασσας. Είναι η πρώτη φορά, αγαπητοί συνάδελφοι, που η Ένωση αναπτύσσει μια ολιστική διατομιακή στρατηγική τέτοιου τύπου που θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη προστασία και προώθηση των συμφερόντων τη Ένωση στον τομέα τη ασφάλεια και τη οικονομία και των κρατών μελών τη όσον αφορά τη θάλασσα. Καθορίζει τα στρατηγικά συμφέροντα και τι απειλέ στον παγκόσμιο στρατηγικό τομέα τη θάλασσα, Προωθεί αρχέ τη Ένωση, ε, το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία, το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια και μια προσέγγιση για την ε, θαλάσσια ασφάλεια που να βασίζεται σε κανόνες όπως εκφράζεται και διεθνή, στο Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα των Ηνωμένων Εθνών. Σε θεσμικό επίπεδο, η έγκριση του κανονισμού για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων είναι επίσης ποιοτικό άλμα για την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία μέσω ουσιοδός Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Και συγχαίρω το Κοινοβούλιο που ενέκρινε αυτό το κείμενο. ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε επίσης στην διεύρυνση, ανενώντας έτσι το ενδιαφέρον της Ένωσης για αυτά και επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση των χωρών αυτών να εκπληρώσουν τα κριτήρια ένταξης. Πριν από μια εβδομάδα χορηγήθηκε καθεστώς υποψήφια χώρα στην Αλβανία, ενώ πριν από πέντε μήνες ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ένταξη με τη Σερβία. Όσον αφορά την Τουρκία, στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης Ένωση-Τουρκία τονίστηκε ότι η πορεία της Τουρκίας προς την Ένωση εξαρτάται από την πλήρωση των υποχρεώσεων της ε, Τουρκίας σε σχέση με την Κύπρο. Όπως ε, ξέρετε, συνολικά η ελληνική προεδρία κατέληξε επιτυχώς 67 νομοθετικά κείμενα και προώθησε άλλα 15 νομοθετικά κείμενα, όπου επετέχθη συνένεση μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου. Αυτό έγινε μόνο σε 4 μήνες, αντί του συνήθους έξα ε, μήνου, λόγω των ευρωεκλογών. Και τα επιτύχαμε με έναν ελάχιστο προπολογισμό, από τον οποίο δαπανίσαμε μόλις 40% τελικά. Τώρα χαιρόμεθα ιδιαίτερα που η νέα Προεδρία, η Ιταλική, θα πάρει τη σκητάλη για να προωθήσει περαιτέρω όλε αυτέ τι πολιτικέ και πρωτοβουλίε. Ε, προσβλέπουμε και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσουν, θα υπερβούν κάθε προσδοκία, του, ώστε το 2014 να θεωρηθεί από όλου ω ένα πολύ επιτυχημένο μεσογειακό έτο. Ένα έτο για το οποίο όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε μπορούν να είναι περήφανοι. Αγαπητοί φίλοι, τις τελευταίες, τις τελευταίες της χρονιές ε, η χώρα μου αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις, αλλά και η Ευρώπη. Πολλοί προέβλεπαν τη λεγόμενη Brexit, δηλαδή ότι η Ελλάδα θα αποχωρούσε από το ευρώ. Ορισμένοι προέβλεπαν ότι ούτε το ευρώ δεν θα επεβίωνε, αλλά το διαψεύσαμε. Λειτουργεί η Ευρώπη. Ναι, μεν η Ένωση μα έχει προβλήματα, αλλά έχει και την ικανότητα να τα επιλύει και να προχωρεί. Αποδείξαμε στους πολίτες μας παντού στην Ένωση ότι μπορούν να συνεργαστούν για να οικοδομήσουν το κοινό τους μέλλον. Βεβαίω, αυτό είναι ευκολότερο σε περιόδου ευημερία, αλλά ακόμη και στι πολύ δύσκολε και επίπονε περιόδου κρίση. Αποδείξαμε ότι οι πολίτε μα όλη την Ευρώπη μπορούν να αλλάξουν τι χώρε του, να τι κάνουν καλύτερε, πιο υγιεί, πιο ανταγωνιστικέ. Ότι μπορούν επιτυχώ να απαιτήσουν αλλαγέ στην ενωσή μα για να γίνει ισχυρότερη, ασφαλέστερη πιο ανταγωνιστική και πιο σταθερή δημοκρατικά. Στι τελευταίε ευρωεκλογέ οι πολίτε μα δεν ψήφισαν κατά τη Ευρώπη. Αντίθετα, ψήφισαν για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Και πιστεύω ότι ήδη έχουμε αρχίσει να ανταποκρινόμεθα. Αλλά πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω από αυτό. Πρέπει η Ένωσή μα να είναι πιο κοντά στι καρδιές των πολιτών μα. Να αποδείξουμε ότι η Ένωσή μα δεν είναι απλώ ένα μάτσο γραφειοκρατικών δικασιών που κανεί δεν παρακολουθεί, δεν καταλαβαίνει ότι είναι κυρίως θέμα των κοινών προοπτικών, των κοινών ιδεωδών που όλοι συμμερίζονται και όλοι αντιλαμβάνονται ευκολότατα. Πριν από 100 χρόνια περίπου ξεκίνησε ένας τρομερά καταστροφικός πόλεμος εδώ και δεν ήταν ο μόνος τις επόμενες περιόδους. Ήταν τρομερός, αλλά δεν ήταν ούτε καν ο πιο τρομερός. Οι λαοί μας υπέφαραν ξανά και ξανά, μία τραγωδία μετά την άλλη για δέκα αιτίες. Τώρα η Ευρώπη είναι όσο ενωμένη ήταν ποτέ, όσο δημοκρατική ποτέ υπήρξε είναι πιο ευημερούσα και πιο σταθερή από ό,τι ήταν εδώ και αιώνες. Όμως οι λαοί μας πρέπει να εμπνέονται από την Ένωση και τις προοπτικές της. Πρέπει να αισθάνονται ότι η Ευρώπη είναι πιο κοντά στις καρδιές τους. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πρώτη και κυριότερη προτεραιότητά σας εδώ στο Κοινοβούλιο της Ένωσης. Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στις καρδιές των πολιτών μας. Γιατί εσείς, εσείς το Ευρωκοινοβούλιο, είστε πραγματικά η καρδιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Τώρα εξ ονόματος Ευρωπαϊκή Επιτροπής ο Πρόεδρος Μπαρόζο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Σαμαρά, αγαπητά μέλη, το τέλος της ελληνικής προεδρίας σημαδεύει επίσης και μια αλλαγή κοινοβουλευτικής περίοδου. Τους τελευταίους μήνες είδαμε ότι ξεκίνησε και η έξοδος από τη βαθύτατη κρίση, την βαθύτερη μάλλον κρίση που ε, έζησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 50. Έχουμε ξεκινήσει τώρα, είμαστε στο δρόμο της ανάκαμψης, αλλά παρόλα αυτά έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Νομίζω ότι είχε σημασία το ότι ακριβώς σε αυτή τη στιγμή μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια από τις χώρες που εφήγησαν περισσότερα από την κρίση, έδειξε ότι είχε την δυνατότητα όχι μόνο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπιζε σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και με πολύ επικοδομητικό τρόπο να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν προσωπικά τον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά για τον τρόπο με τον οποίο αυτός και η ικανότατη ομάδα του προχώρησαν στον τομέα αυτό και ανέλαβαν τις ευθύνες τους και τις ευθύνες του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων χρόνων με την ικανότητα του και την καθοδήγησή του σε δύσκολους τομείς η ελληνική προεδρία έκανε αυτό το οποίο ήταν απαραίτητο οδήγησε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων κάτω από τεράστια χρονική πίεση λόγω και των ευρωπαϊκών εκλογών. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαρά, σε αυτά δεν θα επανέλθω. Αλλά θα ήθελα να σταθώ στα σημαντικά σημεία που έχουν σχέση περισσότερο με την οικονομική κατάσταση. Είναι μια πραγματικότητα ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και βελτιώνεται στην Ευρώπη. 1,6 ανάπτυξη προβλέπεται φέτος και θα φτάσει σε 2% το 2015. Ανεβαίνουν οι επενδύσεις, ε, το συνολικό δημόσιο χρέος μας ε, είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο θα επιθυμούσαμε πριν από την αρχή της κρίσης. Έξι περισσότερες χώρες έχουν βγει από τη διαδικασία υπερβολικού χρέους. Είναι 11 τώρα οι χώρες που εντάσσονται στη διαδικασία αυτή. Ενώ θυμηθείτε ότι το 2011 ήταν 24 οι χώρες κάτω από τη διαδικασία υπερβολικού χρέους. Αυτό δείχνει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πραγματικά λειτουργεί. Τους τελευταίους μήνες και μετά από την επιτυχή έξοδο από τα προγράμματα εποπτείας της Ιρλανδίας ε, και την επιτυχή εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος για τα πιστοτικά ιδρύματα της Ισπανίας ολοκλήρωσε και η Πορτογαλία με επιτυχία τις διαδικασίες. Η κατάσταση στην Ελλάδα και την Κύπρο έχει σταθεροποιηθεί και υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία βελτίωσης ιδιαίτερα σε τομείς όπου υπήρχαν σημαντικές ανισορροπίες. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Σαμαρά και την κυβέρνησή του γιατί έκαναν πραγματικά εξαιρετικές προσπάθειες. Η Ελλάδα μείωσε ακόμα περισσότερο το έλλειμμά της. Έχει διορθώσει επίσης ιστορικά σημεία προβλημάτων και έχει αρχίσει να ανακάμπτει παρά τους προφήτες της καταστροφής η Ελλάδα παρέμεινε ε, μια πλήρης και αφοσιωμένη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θυμίστε ότι τα, πριν λίγο καιρό τα θέματα αυτά τα συζητούσα όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υπήρχαν αυτοί οι οποίοι προέβλεπαν τον Brexit, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι προέβλεπαν την καταστροφή του ευρώ, υπήρχαν ακόμα και αυτοί που προέβλεπαν την πλήρη καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας δεν αρνείται βέβαια ότι η ανάκαμψη είναι άνηση και εύθραυστη. Η ανάπτυξη είναι σε χαμηλά επίπεδα και η ανεργία, ιδιαίτερα η ανεργία των νέων είναι σε υψηλότατα επίπεδα. Δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε να χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Γι' αυτό πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας στις διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται ε, προς επεξεργασία από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή γιατί όπως είπαμε σημειώθηκαν πάρα πολλά θετικά τους τελευταίους μήνες. Κάποιες από τις εξελίξεις αυτές δεν θα τις πιστεύαμε ε, πριν λίγα χρόνια. Αν ρωτούσατε τους αναλυτές πριν λίγα χρόνια, ότι πριν δύο-τρία χρόνια, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τραπεζική ένωση, θα υπήρχε μια εποπτεία απέναντι στις εθνικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλοι έλεγαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε το 2012 τους όρους Τραπεζική Ένωση, δεν δέχτηκαν πολλοί τους όρους αυτούς. Είπαν ότι δεν είναι κάτι τέτοιο ρεαλιστικό. Μιλάτε ε, καλύτερα για δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά όχι Τραπεζική Ένωση. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως υπάρχει και, ο, και οι δύο μηχανισμοί και το Ταμείο για την εξυγίανση των πιστοτικών ιδρυμάτων. Αυτό ήταν ένα σημαντικότατο μήνυμα προς τις αγορές και προς τους πολίτες μας. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι εδώ, είναι σταθερή και θα γίνει αντικείμενο ολοκλήρωσης. Ε, παράλληλα με αυτές τις νομικές ρυθμίσεις αυτό βελτίωσε την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών και την εμπιστοσύνη στις εθνικές οικονομίες. Χωρίς σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρξει η αδίποτε προοπτική ανάπτυξης. Αυτή ακριβώς η προσπάθεια έχει γίνει και μπορούμε να περάσουμε στην ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Έχει υπεράσει πλέον σε ταχύτητα κρουαζιέρας θα έλεγα έχει προχωρήσει δηλαδή αρκετά με σταθερό ρυθμό λόγω ακριβώς και του υψηλού επίπεδου αλληλεξάρτησης των οικονομιών μας. Μετά από τις τελευταίες αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπήρξε μια ομόφωνη θυμίζω ε, συμφωνία γιατί πολλές φορές υπάρχει η άποψη ότι κάποιοι οι οποίοι συμφωνούν στο Συμβούλιο και μετά ξεχνούν τι έχουν συμφωνήσει, αλλά θυμίζω στη συγκεκριμένα η έγκριση των συστάσεων για συγκεκριμένες κάθε φορά χώρες ήταν μια ομόφανη απόφαση βορρά-νότου, δεξιας αριστερά χωρίς διακρίσεις και η διαδικασία αυτή έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου. Βρισκόμαστε τώρα ε, στο πέρασμα από την φάση της κρίσης σε μια προοπτική θετική, μεταρρυθμιστική, στραμμένη στο μέλλον. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς πριν μερικά χρόνια. Αν κάποιος ρωτούσε πριν μερικά χρόνια έχει η δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει τους εθνικούς προϋπολογισμούς πριν υιοθετηθούν, κανένας δεν θα το πίστευε αυτό. Τώρα όχι μόνο κάτι τέτοιο κατέστη εφικτό, αλλά είναι υποχρέωση γιατί ακριβώς η κρίση απέδειξε το πόσον αλληλοεξαρτημένες είναι οι τύχες μας και οι οικονομίες μας. Και αυτό το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν μερικά χρόνια έχει γίνει πλέον πραγματικότητα. Έχει ξεκινήσει μια πραγματική συζήτηση για τις εθνικές οικονομικές πολιτικές και για το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν το σώμα σας, τα κράτη-μέλη και τις κυβερνήσεις για τα επικοδομητικά μέτρα τα οποία έλαβαν και κάτω από τρομερή χρονική πίεση για να εγκρίνουν τις συστάσεις της ειδική αναχώρας στα πλαίσια ε, της ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Πέραν αυτού, δεν είναι σωστό να λέγεται κάτι το οποίο ακούγεται σε ορισμένε χώρε, ότι όλα αυτά τα επιβάλλουν οι Βρυξέλλες, όλα αυτά τα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα πρωτοβουλίας, έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόταση, να ξεκινήσει τη διαδικασία. Είναι και ο αντικειμενικός αν θέλετε διαιτητής ελέγχει αν οι συστάσεις έχουν γίνει αντικείμενο εφαρμογής ή όχι. Αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο από τις κυβερνήσεις και από τους υπουργούς οικονομικών και τέλος από τους πρωθυπουργούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ λοιπόν να μην παρατείνουμε μια τέτοια παρανόηση γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις και πρέπει να έχουν όλοι το θάρρος να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Τώρα, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα θέματα της εφαρμογής. Δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί. Απαιτούνται περισσότερες αλλαγές, περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στην απασχόληση, τις εγγυήσει για τους νέους, στην καταπολέμηση του αποκλεισμού του κοινωνικού κτλ. Αυτές είναι από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που συνέβησαν τους τελευταίους έξι μήνες. Το ευρωπαϊκό λοιπόν εξάμεινο και η ολοκλήρωση της διαδικασίας που οδήγησε στην τραπεζική ενότητα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομείς, στους οποίους θα πρέπει επίσης να επιταχύνουμε. Και η επερχόμενη Προεδρία έχει πολλά να κάνει έτσι ώστε να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες δράσεις στην καταπολέμηση κυρίως της ανεργίας των νέων. Πρέπει λοιπόν εμείς να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, από τους προϋπολογισμούς μας τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για, Marshall, για σχέδιο Marshall για την Ευρώπη. Ο προπολογισμό μα είναι πολύ μεγαλύτερο για τα επόμενα 7 χρόνια. Αν τα χρήματα που θα έχουμε στη διάθεσή μα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επόμενα 7 χρόνια χρησιμοποιηθούν σωστά και με σωστέ επενδυτικέ δυνατότητε, τότε θα ωφεληθούν πάρα πολλοί οι χώρε που δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν τι απαιτούμενε διορθώσει μόνε του. Ε, τα αποτελέσματα και σε σχέση με το Refit ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι αποφάσεις. Ε, τα τελευταία έξι μήνες μέσω του προγράμματος REFIT έχουμε κάνει πάρα πολλές νομοθετικές αλλαγές χρήσιμες. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Ήδη από το 2006 έχουμε αποσύρει πάρα πολλές ρυθμίσεις ε, νομικές που ίσχυαν δεν γίνεται γνωστό αυτό για να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Πολλοί μιλούν για την γραφειοκρατία που επιβάλλεται από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όλε οι κυβερνήσει έκαναν την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε θα είχε δημιουργηθεί ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον για τους συμπολίτε μας και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι το 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού γίνεται αντικείμενο διαχείρισης από τα ίδια τα κράτη-μέλη και το 1 τρίτο ε, προέρχεται από τις πράξεις εθνικής εφαρμογής των κοινοτικών αποφάσεων. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο να είναι λιγότερο γραφειοκρατικό, ένα περιβάλλον το οποίο να είναι φιλικό προς την ανάπτυξη και σε αυτό θα βοηθήσει και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε συζητήσει και άλλα θέματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Δεν θα ήθελα να σταθώ τώρα λεπτομερώς σε τομείς όπως ε, η δικαιοσύνη, η ελευθερία ε, και ασφάλεια, ιδιαίτερα η μετανάστευση. Και τέλος να πω δύο λόγια γι' αυτό. Διότι δέκα χρόνια μετά τη μεγάλη διεύρυνση του 2004, τι συμβαίνει. Ας μην ξεχνάμε, το 2004 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρώτη μου Επιτροπή ανέλαβε τα ενία, βρισκόμαστε στις αρχές του 2004 μόνο 15 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα είμαστε 28, σχεδόν διπλασιάστηκαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ιστορικά όσον αφορά την ευρωπαϊκή ιστορία, ότι επανενώθηκε η Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό <clears throat> θα πρέπει να το θυμόμαστε το 2014 αυτό διότι 25 χρόνια μετά την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος, 70 χρόνια μετά την απόβαση στη Νορμανδία και 100 χρόνια μετά το τέλος, την έναρξη του ε, Πρώτου Ευρωπαϊκού Πολέμου. Ε, εορτάζουμε την επανένωση της Ευρώπης και βλέπουμε ότι είναι ανοιχτή προς το μέλλον αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνενώνει πιο πλούσια και λιγότερο πλούσια κράτη παλαιότερα και νεότερα, βόρα και νότο, ανατολή και δύση. Αυτά τα κράτη-μέλη έγιναν ισχυρότερα, οικονομικά, πολιτικά, δημοκρατικά από το 2015 βλέπουμε ότι η ε, Λετωνία ε, εντάσσεται στο ευρώ. Η Λιθουανία θα είναι το 19ο κράτος μέλος ε, το 2015 της Νομισματικής Ένωσης. Ένα κράτος που πλούτος του αυξήθηκε από το 35% του μέσου όρου του ΑΕΠ, του κοινοτικού ε, ε, ΑΕΠ, ε, στο 75% αυτού του μέσου όρου του κοινοτικού ΑΕΠ. Πώς μπορούν να είναι αρνητικοί λοιπόν οι πολίτες όσον αφορά την διεύρυνση και την ενοποίηση της Ευρώπης. Πώς είναι δυνατόν να μην κατανοούν τη μεγάλη μηχανή ολοκλήρωσης, δημιουργίας ευκαιριών που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εργαζόμαστε ώστε να υπάρξει η σταθεροποίηση, η σταθερότητα, αποφεύγοντας τη δημιουργία ε, ουκρανικών περιπτώσεων γύρω από την Ευρώπη, διότι αυτό θα συνέβαινε αν δεν είχε επιτευχθεί η διεύρυνση. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ανοιχτή η Ευρώπη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήταν μεγάλο σφάλμα να πει κανεί ότι θα κλείσουμε τα σύνορά μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προκλήσεις, σίγουρα ναι, αλλά πρέπει με βάση αρχέ ε, να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάχρηση των δικαιωμάτων ελευθερίας κυκλοφορία. αλλά θα ήταν μεγάλο σφάλμα για την Ευρώπη να κλείσουμε, να στεγανοποιήσουμε τα σύνορά μα. Το βλέπουμε αυτό. Και σε σχέση με την Αλβανία η πρόοδος ε, που ε, γίνεται θα ε, βοηθήσει να μας προσεγγίσει. Θα ήταν λοιπόν πολύ ανεύθυνο πράγμα να μην υπάρξει ελπίδα για αυτές τις χώρες αν υλοποιούν συγκεκριμένες, ε, ε, συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα είναι όριμες. Ήταν λοιπόν ε, μια τρικυμιώδης περίοδος και δύσκολες οι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν και από πλευράς του Πρωθυπουργού Σαμαρά έγινε αυτό και υπάρχει επίσης και οι μεγάλοι, υπάρχουν επίσης οι μεγάλες εθνικές παραδόσεις. Παραδόσεις που ήταν και παρούσες κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας και μπορούν να περιγραφούν με τρεις ελληνικούς όρους ε, που προσεγγίζουν την ευρωπαϊκή μας προσέγγιση όσον αφορά τον ε, λόγο, λόγο, τον ορθό λόγο δηλαδή και το ορθό για την Ευρώπη το πάθος, ακούγοντας δηλαδή και κατανοώντας όλες τις πλευρές και τα αιτήματα των πολιτών μας και το ήθος ήθος όσον αφορά την διασφάλιση των ευρωπαϊκών αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρόζο. Κυρίε και κύριοι, πρωτού ξεκινήσει η συζήτηση τώρα με την ημερήσια διάταξή μας έχουμε σχεδόν 35-40 λεπτά καθυστέρηση. Και γι' αυτό τώρα την εκλογή των κοσμητόρων δεν θα την καθορίσουμε για τις 12 ε, και 35 αλλά για τις 13.00 ε, η ώρα. Θα ήμουν ευγνώμων αν αυτό θα μπορούσε να αναφερθεί και να αντανακλάται και στις οθόνες ώστε να το ξαναπούμε ότι η εκλογή των κοσμητώρων δεν θα γίνει στις 12.30 όπως προβλεπόταν, αλλά στις 1, η ώρα. Αν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε πιο πριν τη συζήτηση, πριν από τη μία η ώρα, τότε θα γίνει η εκλογή των κοσμητόρων νωρίτερα. Αλλά θα συνεχίσουμε μέχρι μία η ώρα. Και περνάμε τώρα και έχει τον λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚΑ ο κύριος Κεφαλογιάννης. Παρακαλώ κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη από την ίδρυσή της κάνει πάντα δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω αλλά πάντα υπάρχει ένα βήμα μπροστά για να προχωρούμε στην ευρώπη της ανάπτυξης της αλληλεγγύης στην ευρώπη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε παρά τις αντίξωες συνθήκες σε ελλάδα και ευρώπη η ελληνική προεδρία για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης με την υιοθέτηση του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης με την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης υιοθετώντας οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των δημοσίων προμηθειών για το e banking για το e commerce για την πάταξη της φοροδιαφυγής με την προώθηση του τομέα της μετανάστευσης με υιοθέτηση των οδηγιών για την ενδοεπιχειρησιακή μετακίνηση προς τρίτες χώρες μειοθέτηση του κανονισμού για τη frontex. είναι αλήθεια αυτό που είπε ο πρωθυπουργό ότι μόνο σε τέσσερις μήνες η ελληνική προεδρία ολοκλήρωσε 67 νομοθετικά κείμενα. πέτυχε συνένεση με το συμβούλιο σε 15 νομοθετικά άλλα κείμενα για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος για την τρομοκρατία για την europol για την προστασία των παιδιών σε ποινικέ διαδικασίες. με την προώθηση πολιτικών για την Ελληνική με την υιοθέτηση του κανονισμού για το ευρωπαϊκό ταμείο αλληλεγγύης για τις φυσικές καταστροφές με τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση των φακέλων για τη διεύρυνση σε αλβανία μαυροβούνιο και σερβία με την προώθηση της διαφάνειας με τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τις επιχειρήσεις. κύριε πρόεδρε η ιταλική προεδρία παίρνει τώρα τη σκητάλη ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ιταλική προεδρία συγχαίρομαι την ελληνική προεδρία που πήγε μπροστά τα πράγματα για την ευρώπη γιατί η λύση στην ευρώπη είναι η διεύρυνση και η ευάθυνση των δημοκρατικών θεσμών όχι ο λαϊκισμός όχι ο ευρωσκεπτικισμός. σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. αγαπητέ πρόεδρε και πρωθυπουργέ της ελλάδος η παράταξή μου συμμετέχει στην κυβερνητική συνεργασία στην ελλάδα και εν μέσω μιας ομολογουμένως επιτυχημένης προεδρίας που όντως έβαλε προτεραιότητα την στήριξη των νέων των ανέργων την ανάπτυξη αλλά και την ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης όπως είπε και ο κύριος μπαρόζο που θα αντιμετωπίζει ισότιμα όλες τις χώρες μέλη. πήραμε και τα μηνύματα των ευρωεκλογών και οι έλληνες λοιπόν ζήτησαν ευρύτερες πολιτικές συμμαχίες αλλά και περισσότερη ευρώπη και αυτό παρά τις λανθασμένες επιλογές του ευρωπαϊκού συμβουλίου και τα στρατηγικά λάθη για σκληρή λιτότητα που έφερε ανάμεσά μας και ευρωσκεπτικιστές αλλά και ακροδεξιούς. η ευρωπαϊκή ένωση όφιλε να επιλέξει ή έστω να εφεύρει έναν άλλο δρόμο για να μπορούμε να μιλάμε για την επιτυχία της ευρώπης της αλληλεγγύης καθώς η ελλάδα ό,τι πέτυχε το πέτυχε με σκληρές θυσίες των ελλήνων και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας καθώς βρεθήκαμε απροετοίμαστοι να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους ευρωπαίους πολίτες. ας ελπίσουμε πως ε, η ελληνική η ιταλική προεδρία που ακολουθεί την ελληνική θα συνεχίσει την προσπάθειά μας για την έβρεση ενός άλλου δρόμου με ευαισθησία αλλά και ευελιξία στην εφαρμογή του συμφώνου και την επαναφορά φυσικά των κόκκινων γραμμών όπου αυτές παραβιάστηκαν γιατί δεν είναι πια αυτονόητα όσα θεωρούσαμε ότι είναι. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Καηλή. Τώρα θα λάβει τον λόγο για την ECR ο κύριος Νότης Μαριάς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως αντιπρόεδρος του ECR της κατεξοχήν αντιφεδεραλιστικής πολιτικής ομάδας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ελληνική προεδρία είναι ένα μνημείο αποτυχίας. δεν πρόκειται βέβαια για κανένα success story όπως δεν πρόκειται και για success story σε σχέση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει στην πατρίδα μας την ελλάδα μια μνημονιακή πολιτική η οποία έχει διαλύσει τη χώρα. κύριε πρόεδρε από το μάιο του 2010 μέχρι σήμερα η ελλάδα έχει πάρει 214 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια ένα τεράστιο ποσό πάνω από το 120% του αεπ και θα φανταζόταν κανείς ότι με αυτό το ποσό θα μπορούσε να είχε αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία να είχε απογειωθεί. ποια είναι όμως η πραγματικότητα; 1,5 εκατομμύριο άνεργοι χιλιάδες μαγαζιά κλειστά 6.000 χιλιάδες αυτοκτονίες σαράντα μείωση των μισθών και των συντάξεων 40% του ελληνικού πληθυσμού κάτω από τα όρια της φτώχειας το 175% πλέον του αεπ ανέρχεται το δημόσιο χρέος δημοσιονομικό έλλειμμα 11,5% psi με το οποίο διαλύθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ για να σωθούν οι έλληνες ολιγάρχες οι οποίοι ήταν οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών. η ελλάδα λοιπόν μετατράπηκε σε κοινωνικό νεκροταφείο γιατί ο κύριος σαμαράς ακολούθησε την πολιτική της τρόικας. χάσατε την ευκαιρία κύριε σαμαρά να θέσετε όλα εκείνα τα θέματα που για δεκαετίες απασχολούν την ελλάδα και η διεκδίκησή τους εκτός από ιστορική επιταγή είναι και άμεσης ζωτικής σημασίας για την οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας. χάσατε την ευκαιρία να ταυτιστείτε μαζί με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ενάντια στην τρόικα ενώ εσείς στηρίξατε την τρόικα. χάσατε την ευκαιρία να σταματήσει η πολιτική της λιτότητας την οποία εσείς στηρίξατε ως κλασικά μερκελική πολιτική. χάσατε την ευκαιρία να ανακαλέσετε στην τάξη την επιτροπή η οποία υπηρετεί τους δανειστές χάσατε την ευκαιρία να καλέσετε τον κύριο ντράγκη και την παρέα του να μην κερδοσκοπεί σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού πληρώνοντας ο ελληνικός λαός στο 100% τα ομόλογα που αγόρασε η κεντρική τράπεζα με έκπτωση τουλάχιστον. 40%. μνημείο λοιπόν αποτυχίας η πολιτική σας στην ελλάδα αλλά και σε επίπεδο προεδρίας της ευρωπαϊκής ένωσης. Τώρα θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ε, Ενωτικής Αριστεράς η κυρία Σακοράφα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς η συνθήκη της Λισαβόνας αποδυνάμεσο το ρόλο της εκπεριτροπής Προεδρίας ώστε τελικά η προεδρεύουσα χώρα να καλείται να υλοποιήσει προηλημμένες αποφάσεις από τεχνοκράτες και εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες που μετέχουν στα διακυβερνητικά όργανα. Για ποιον λοιπόν είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη μια προεδρία? Τα ευρωπαϊκά διευθυντήρια μιλάνε για εντυπωσιακή δουλειά, εξαιρετικά αποτελέσματα και συνετή, σπαρτιατική σχεδόν οικονομική διαχείριση και μάλιστα για αυτό που στην αρχή τη ε, ανάληψη τη Προεδρία τον ανέφεραν σαν τον πλέον αδύναμο κρίκο. Αυτό για μας σημαίνει ότι η ελληνική προεδρία ακολούθησε πιστά την νεοφιλελεύθερη πολιτική άκρα της λιτότητας χωρίς να θέσει το παραμικρό ανάγχωμα παρά τα τρανταχτά επιχειρήματα που είχε δεδομένης της πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα και μάλιστα στην καρδιά της ευρώπης. και αυτό είναι απειλή για όλους τους λαούς της ευρώπης μιας και η ελλάδα είναι πιλότος για όλα όσα θέλουν να εφαρμόσουν και θα αναφερθώ σε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα κατάργηση των συλλογικών ε, ε, διαπραγματεύσεων πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων παντελή απουσία του κράτους από δαπάνε για υγεία συντάξεις κοινωνικές παροχές και πρόνοια πλήρη απελευθέρωση της ασίδωτης δράση των μεγάλων μονοπωλίων ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στο όνομα της αποπληρωμής ενός μεγάλου χρέους ενός χρέους το οποίο ποτέ δεν ελέγχθηκε και φορτώθηκε ο ελληνικός λαός. σε θέματα δε κυρίαρχης πολιτικής όπως η τραπεζική ένωση η δημοσιονομική εξυγίανση οι μηχανισμοί οικονομικής διακυβέρνηση και άλλα η απουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων ήταν κραυγαλαία θα κλείσω με δύο άκρως σημαντικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας που καταδεικνύουν ότι η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης αποφασίζεται ερήμην των κυβερνήσεων των κρατών μελών των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και του ίδιου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και αυτό είναι κυρίαρχο θέμα δημοκρατίας και μας αφορά όλους. αναφέρομαι στην ουκρανική κρίση και στο ζήτημα των χημικών της συρίας και στι δύο περιπτώσει, τα οικονομικά συμφέροντα ήταν αυτά που καθόρισαν σε απόλυτο βαθμό την πολιτική συμπεριφορά των κυβερνήσεων που στηρίζουν. για μα, μια τέτοια επιτυχημένη προεδρία αποδείχθηκε καταστροφική για τον ελληνικό λαό συνιστά απειλή για του λαού τη Ευρώπη και είναι επικίνδυνη για το μέλλον της ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. δεσμευόμαστε από κοινού με τους ιταλούς μας να αγωνιστούμε ώστε η ιταλική προεδρία να μην έχει τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τον λόγο τώρα θα λάβει εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων ο κύριος, για τους Πράσινους ο κύριος Γκίγκολτ. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Σαμαρά, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι είμαι απογοητευμένος. Δεν είμαι Έλληνας, αισθάνομαι ότι είμαι ξένος σε αυτή τη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα δύο λόγια να πω και να αποσαφηνίσω σε σχέση με το τελευταίο εξάμεινο και την ε, ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την ολοκλήρωση μια ολόκληρη σειρά χαρτοφυλακίων που είναι πολύ σημαντικά για τη σταθερότητα των οικονομικών αγορών και φυσικά και για την Τραπεζική Ένωση. Η Τραπεζική Ένωση είναι το μεγαλύτερο βήμα για τη σταθεροποίηση του ευρωπαϊκού οικονομικού Συστήματο. και προ αυτή την κατεύθυνση κάναμε ένα μεγάλο βήμα για την Ευρώπη προ τα εμπρό. Με ανησυχία βλέπω τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το έργο της ότι στο μέλλον τα ε, ταμεία διάσωσης θα πρέπει από τις μικρές ε, ε, τράπεζες να χρηματοδοτείται το ταμείο αυτό υπερβολικά σε ποσοστό από τις μικρές τράπεζες και όχι αναλογικά όπως θα έπρεπε από τις μεγαλύτερες τράπεζες. Θα πρέπει για την Ευρωζώνη μια, μια ολόκληρη σειρά έτρων να εμβαθυνθεί. Για την Τραπεζική Ένωση είναι ένα μεγάλο σχέδιο που το έχουμε συζητήσει θέματα των ε, προεδριών, των τεσσάρων προεδριών και προτάσεις. Ε, δεν έγιναν πολλά από αυτά. Ήταν μια πολιτική που ακολουθούσε μια μονόπλευρη λιτότητα και υπήρχε και ένας επιθετικός ε, ανταγωνισμός φορολογικός. Δεν έγιναν πολλά πράγματα για τις επενδύσεις. Έχουμε μεγάλη ανεργία και έχουμε ελλειπή δίκαια χρηματοδότηση και γι' αυτό γίνεται λόγος τώρα και για νέα χρέη. Με αυτόν τον τρόπο η άδικη χρηματοδότηση, η φοροαποφυγή, ο φοροανταγωνισμός, λίγα πράγματα έκανε η Προεδρία σχετικά και ελπίζω ότι το επόμενο εξάμεινο θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια εξ ονόματος ε, <clears throat> των μη εγγεγραμμένων ο κύριος Επιτίδιος παρακαλώ. Πριν από λίγο ο κύριος Μπαρόζο ομίλησε και είπε ότι τώρα η ευρώπη είναι περισσότερο ενωμένη και περισσότερο δημοκρατική. όλοι γνωρίζετε ότι η αρχαία ελλάδα υπήρξε το λίκνο της δημοκρατίας. εκείνο που ίσως πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε είναι ότι στη σύγχρονη ελλάδα την ώρα που ο ελληνικός λαός υφίσταται τις συνέπειες εφαρμογής των μνημονίων της τρόικα δηλαδή οικονομική εξαθλίωση πείνα φτώχεια ανεργία αβάστακτη φορολογία και αυτοκτονίες πολιτών μια ολιγαρχική συγκυβέρνηση των κυρίων σαμαρά και βενιζέλου των επικεφαλής δηλαδή του δευτέρου και τετάρτου σε εκλογική δύναμη πολιτικών κομμάτων όπως απέδειξαν οι πρόσφατες ευρωεκλογές έχει καταργήσει τη διάκριση των εξουσιών η οποία είναι βασική αρχή της δημοκρατίας. χειραγωγώντας τη δικαιοσύνη και παρεμβαίνοντας στο έργο της έχει καταστρατηγήσει θεμελιώδεις αρχές του συντάγματος της χώρας μας. συγκεκριμένα προκειμένου να εξουδετερώσει τον ουσιαστικό και μοναδικό πολιτικό της αντίπαλο το κόμμα της χρυσής αυγής την τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας επειδή δεν έχει πολιτικά επιχειρήματα για να το αντιμετωπίσει φυλάκισε τον αρχηγό του και έξι από τους βουλευτές χωρίς να αποδεικνύονται εναντίον τους κατηγορίες σε όσους δεν έχει φυλακίσει απαγορεύει να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του κόμματος. η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη διότι προσβάλλει τις αρχές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. για τον λόγο αυτό ο κύριος σαμαράς όφιλε παράλληλα με τον απολογισμό των πεπραγμένων της ελληνικής προεδρίας να απολογηθεί ενώπιόν σας για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κυβέρνησής του. Ζητούμε από εσά και ολόκληρο το πολιτικό ε, δημοκρατικό κόσμο τη Ευρώπη να καταδικάσει τι παράνομε πρακτικέ τη ελληνική κυβερνήσεω. Επιδίωξή μα είναι να σταματήσει η παράνομη πολιτική δίωξη και να αποφυλακιστούν. Σα ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε, σα ευχαριστούμε. Ξεπεράσατε κατά πολύ το χρόνο σα, σα ευχαριστούμε. Τώρα για το ΕΛΚ θα... λάβει τον λόγο η κυρία Σούικα. Ελπίζω ότι σωστά πρόφερα το όνομά σα. Κυρία Σούικα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είδα ότι ζήτησαν να παρέμβουν περισσότερο Έλληνες συνάδελφοι Ευρωβουλευτές και εμπλέκονται σε συζητήσεις για τα εσωτερικά της Ελλάδας, για εσωτερικά πολιτικά θέματα της Ελλάδας. Εγώ όμως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαμαράκη ονόματος της Ελληνικής Προεδρίας για όλες τις προσπάθειες κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας που έγιναν παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα κατά την περίοδο της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Σαμαρά θερμά. Έλαβα τον λόγο <clears throat> και σε σχέση και με την παρουσίαση των δικών σας προτεραιοτήτων θα ήθελα να παρέμβω και να πω και πάλι ότι χαίρομαι ότι θέτεται κέντρο βάρους στην ε, θαλάσσια πολιτική και ναυτιλιακή πολιτική και σε σχέση με την ε, περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής ε, παρουσιάζοντας και τα αποτελέσματα της ελληνικής προεδρίας. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια μεγάλη πολιτική επιτυχία αυτή και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό το έργο στο μέλλον. Όταν έχουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Προεδρίας σας που αναφέρθηκαν, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι αυτά τα οποία συνέβησαν όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, τα οικονομικά θέματα και τον ενιαίο μηχανισμό αντιμετώπισης ε, προβλημάτων, θα ήθελα να πω ότι ήταν και αυτά επιτυχή. Η αντιμετώπιση όμως της ανεργίας και της ανεργίας των νέων παραμένει πρόβλημα. Συμφωνώ με τον πρόεδρο Μπαρόζο που είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί το έργο μας κατά της ανεργίας και τη ανεργία των νέων. Έχουμε μια ολόκληρη σειρά μέσων ως Ευρώπη στη διάθεσή μας που δεν τα είχαμε κατά το παρελθόν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα και κατά την Ιταλική Προεδρία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια ο κύριος Κύρκος παρακαλώ εξ ονόματος των SD. Κύριε Πρωθυπουργέ, επιτυχημένη ή διαχειριστική η πέμπτη ελληνική Προεδρία από τη μια μεριά, η Προεδρία συνέχισε όλα τα ζητήματα τη κοινοτική νομοθεσία που ήταν σε εξέλιξη. Σε μερικά δε από αυτά επήλθε συμφωνία σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η πολιτική συμφωνία για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανση και το ταμείο του και στη θαλάσσια πολιτική η συμπερίληψη αναφορά για το σεβασμό στο δίκαιο τη θάλασσα. από την άλλη όμω, η προεδρία δεν πήρε τι απαραίτητε πρωτοβουλίε σε θέματα που είχε θέσει η ίδια ως προτεραιότητε όπως το θέμα τη ανεργίας των νέων που τείνει να εξελιχθεί σε δομικό στοιχείο των κοινωνιών σε κρίση και στο μεταναστευτικό ζήτημα όπου περισσότερη αλλαγή στην πράξη είναι απαραίτητη εκ μέρου τη Ένωση σα προτείνω κύριε πρωθυπουργέ να συνεργαστείτε στενά με την επερχόμενη ιταλική προεδρία για την ουσιαστική αντιμετώπιση του κοινού προβλήματο. και ενώ δεν είδαμε συγκεκριμένε προτάσει σε καυτά ζητήματα η προεδρία προώθησε το αμφιλεγόμενο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών παρέχοντα περισσότερα δικαιώματα στι πολυεθνικέ εταιρείε. ακόμα απορούμε γιατί. εντελώ απούσα ήταν η προεδρία στο πρόβλημα τη Ουκρανία, ενώ τα άλλα θεσμικά όργανα βρίσκονταν επί τέλο από μια χώρα που λειτουργήσε ω πειραματόζωο για την αντιμετώπιση τεράστια κρίση θα περίμενε κανεί να ληφθούν πρωτοβουλίε ώστε να ενισχυθεί η κοινοτική μέθοδο και η δημοκρατία στη σχέση ευρωπαϊκή επιτροπή και κρατών μελών. δυστυχώ δεν είδαμε κάτι τέτοιο. η ελληνική προεδρία προσπάθησε με σοβαρότητα όμω δεν άγγιξε του στόχου που ίδια είχε θέσει ίσω γιατί επικεντρώθηκε στην πιο γραφειοκρατική αν και αναγκαία δουλειά. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κύρκο. Επόμενος ε, για ένα λεπτό ο συνάδελφος κύριος Παπαδάκης παρακαλώ. Μικρό. Μικρόφωνο παρακαλώ. Την αντιλαϊκή αποστολή που είχε αναλάβει προώθησε περαιτέρω την αντιλαϊκή πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης καταφέρνοντας νέα πλήγματα στα δικαιώματα των εργαζομένων στην ελλάδα και σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ενίσχυσε το μεγάλο κεφάλαιο στα πλαίσια της νέας οικονομικής διακυβέρνησης και της λεγόμενης τραπεζικής ένωσης στρεφόμενη κατά των λαών. η συγκυβέρνηση νέας δημοκρατίας και πασόκ ανέλαβε δραστήριο ρόλο για λογαριασμό της ελληνικής αστικής τάξης στην προώθηση της υπερρεαλιστικής στρατηγικής και το σχεδιασμό της ευρωπαϊκής ένωσης πρωτοστάτησε στην ανοιχτή υπερρεαλιστική επέμβαση ευρωπαϊκής ένωσης ηπα και νατο στην ουκρανία στη στήριξη της κυβέρνησης των φασιστικών δυνάμεων εκεί διέθεσε το ευρωνοσιακό στρατηγείο στην ελλάδα για τη διεύθυνση της υπεριαλιστικής στρατιωτικής επέμβασης της ευρωπαϊκής ένωσης στην κεντροαφρικανική δημοκρατία προώθησε τη στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας της ευρωπαϊκής ένωσης για τη συγκρότηση ναυτικής πολεμικής δύναμης πυρός της ευρωπαϊκής ένωσης ενάντια στους λαούς απέναντι σε αυτή την ενιαία επίθεση ενιαία πρέπει να είναι και η πάλη των λαών. το κομμουνιστικό κόμμα της ελλάδας θα παλέψει για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Παπαδάκη. Ακολουθεί για 1,5 λεπτό ο κύριος Κεφαλογιάννης. Παρακαλώ. Τρεις παρατηρήσεις πρώτον θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους και ιδιαίτερα από την ελλάδα ότι βρισκόμαστε στο στρασβούργο δεν βρισκόμαστε στην αθήνα. μπορούμε να διοργανώσουμε μια ημερίδα να συζητήσουμε τα θέματα του εσωτερικού της ελλάδος. παρατήρηση δεύτερη έχει πολύ δίκιο που στο πρώτο σύνθημα που είχαμε σε ευρωεκλογές στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα ήταν η μάχη εναντίον του λαϊκισμού. αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα τη δώσουμε ενάντια στους λαϊκιστές και θα προχωρήσω με τις ιδέες της ευρωπαϊκής ένωσης αυτές που οδηγούν στην ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. παρατήρηση τρίτη η λύση στην ευρώπη είναι περισσότερη ευρώπη είναι καλύτερη ευρώπη είναι διεύρυνση και εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών και αυτός είναι ο στόχος μας. και μια παρατήρηση κύριε πρόεδρε που αφορά την κρίση αν η ευρώπη βίωσε την κρίση τόσο δραματικά είναι γιατί δεν είχε τα εργαλεία αν συγκρίνουμε την ευρώπη με τις ηνωμένες πολιτείες οι ηνωμένες πολιτείες διαχειρίζονται το 6% του ακαθάριστου εθνικού τους προϊόντος σε ομοσπονδιακό επίπεδο εμείς το ένα οι ηνωμένες πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν ομόλογα εμείς δεν μπορούμε και στην περίοδο της κρίσεως τύπωσαν χρήμα έστω και λίγο πληθωριστικό σε 7 τράπεζες. εμείς λοιπόν πρέπει να δούμε το ευρωπαϊκό όραμα την περισσότερη ευρώπη την καλύτερη ευρώπη να πάμε μπροστά η ειρήνη η οποία κατοχυρώθηκε τα προηγούμενα 60 χρόνια οφείλεται στον ευρωπαϊκό οραματισμό και η παγίωση της δημοκρατίας στις νότιες χώρες της ευρώπης και τώρα στις ανατολικές χώρες της ευρώπης οφείλεται στο ευρωπαϊκό όραμα και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Κεφαλογιάννη. Ακολουθεί για ένα λεπτό συνάδελφος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Σαμαρά και τον πρόεδρο Μπαρόζο. Είπαν ότι οι γενναίες που ε, ακολουθούν και με βάση αυτά που κάναμε θα έχουν πολύ σημαντικά επιτεύγματα στη διάθεσή τους. Εδώ και πάνω από 50 χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε τώρα μεγάλες αλλαγές που έχουμε επιτύχει. Εδώ και 70 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια, εδώ και 10 χρόνια όλα όσα επιτύχαμε είναι μεγάλα επιτεύγματα. Όμως οι νέοι οι νέοι που είναι 20-25 ετών δεν θέλουν να ακούν για αυτά τα επιτεύγματα. Θέλουν να ακούν για τη συζήτηση για το, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για την ανεργία, την ε, αδικία, τα προβλήματα που δεν επιλύονται στη ζωή τους. Και λένε χάνουμε την πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνουν την πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα νέο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να ξεκινήσει και πάλι μια νέα κίνηση να έχει η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Λιβεράσκη. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Έχετε εσείς τον λόγο κύριε Πλέκοβιτς παρακαλώ. E, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά για την αναλυτικότατη παρουσίασή του. Ενθυμούμε το 2003 ότι είχαμε συναντηθεί όταν η ε, χώρα μου, η Κροατία, είχε υποβάλει την αίτηση ένταξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συγχαρώ την Ελληνική Προεδρία και τον Πρωθυπουργό και για την πολιτική στον τομέα της θάλασσας, όπως επίσης και για τις συγκεκριμένες πολιτικές στην, ε, για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιωνίου Πελάγους. Είναι μια περιοχή σημαντική. Σας συγχαίρω επίσης και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την Τραπεζική Ένωση, όπως επίσης και για το θέμα του καθεστώτος λειτουργίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε Πλένκοβιτς. Ακολουθεί ο συνάδελφος Μάντρετς, παρακαλώ. Herr ο κύριος Μαυρίδης παρακαλώ. Συνάδελφε Μαυρίδη, έχετε τον λόγο. Θέλω και, <clears throat> θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας για τα επιτεύγματα που έχουν γίνει μέσα από τέτοιες δυσκολίες παρόλο που ομολογουμένως έχουν γίνει και λάθη σε αυτή την πορεία. Όμως θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο το οποίο αφορά και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου το θέμα των απειλών και το θέμα της ασφάλειας της θάλασσας το οποίο φυσικά έχει να κάνει με την ενέργεια και φυσικά αυτό αφορά ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση. θεωρώ λοιπόν ότι τα μικρά κράτη τα οποία είμαστε ενταγμένα στην ευρωπαϊκή ένωση προσδοκούμε στη στήριξη της ευρωπαϊκής ένωσης για να μπορέσουμε να ασκήσουμε το κυρίαρχο δικαίωμά μας να αξιοποιήσουμε την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη για το συμφέρον των λαών μας αλλά και για το συμφέρον της ίδιας της ευρωπαϊκής ένωσης. και τέλος χαιρετίζω ένα σημείο ότι η όποια πορεία της τουρκίας προς την ευρωπαϊκή ένωση δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε βήμα χωρίς την αποδοχή των αρχών της ευρωπαϊκής ένωσης και της κύπρο. ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Μαυρίδη. Η κυρία Θεοχάρου, παρακαλώ τώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη διάρκεια του Συμβουλίου Σύνδεσης της Τουρκίας ε, παρέδωσε στον, Υπουργό Εξωτερικών Βενιζέλο έγγραφο 64 σελίδων στο οποίο αναφέρεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υφίσταται πλέον, είναι κλινικά νεκρό ποια ήταν η εκδήλωση αλληλεγγύης εκ μέρου της ευρωπαϊκής ένωσης προς ένα κράτος μέλος το οποίο ε, ε, θεωρείται κλινικά νεκρό από ένα, κράτος μέλος, ε, που διεκδικεί την ένταξή του και πώς αντέβρασε η ελλαδική προεδρία όταν η τουρκία καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου ζήτησε την αναγραφή του τίτλου ε, ελληνοκυπριακή διοίκηση στα διαβατήρια εκείνων που ετούνται αίτηση εισόδου στην ε, Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία συνάδελφε Θεοχάρος. Ο κύριος συνάδελφος Ντενάνο παρακαλώ. Συνάδελφε Ντενάνο παρακαλώ. Okay, möchte nicht sprechen. Δεν θέλει να παρέμβει, εντάξει. Η κυρία Γκάλπερτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρωθυπουργέ, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας επενέσω εσάς και την Προεδρία σας για το έργο που επιτελέσατε. Στο έργο σας επικεντρωθήκατε στην οικονομική ανάπτυξη, το, την ανταγωνιστικότητα, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σωστή αυτή η προσέγγιση και επικέντρωση και είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνει η Ευρώπη για το μέλλον. Μου φαίνεται ότι έχετε ε, στέψει με επιτυχία αυτές τις πρωτοβουλίες σας και μπορείτε να είσαστε υπερήφανος για όσα επετέφθησαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Να αναφέρω όμως ε, κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα, το θέμα της ανεργίας των νέων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ανεργίας των νέων και να βελτιωθούν οι προοπτικές για τους νέους. Και γι' αυτό λοιπόν το σχέδιο εγγύησης ε, για τους νέους είναι πολύ σημαντικό και για την Τραπεζική Ένωση. Και αυτό το θέμα έχει τεράστια σημασία και πρέπει να συνεχίσουμε το έργο προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποια χαρτοφυλάκια που παραμένουν ανοιχτά, δεν επετεύχθη επαρκή πρόοδο επ' αυτών. Για παράδειγμα, θέματα ενία αγορά. Όμω, παρόλα αυτά, συνολικά ήταν πολύ ικανοποιητικό το έργο σα και σα συγχαίρω γι' αυτό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφο Ντενάνο, τώρα θέλει να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Δεν είχα ζητήσει το λόγο, αλλά μιας και μου το δώσατε, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Καταρχά θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου απέναντι στον ελληνικό λαό, τον οποίο γνωρίζω γιατί έχω ζήσει αρκετά στη χώρα αυτή. Οι Έλληνες ήταν πάντα ιδιαίτερα λέει, και γι' αυτό πέρασαν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και θέλω να χαιρετήσω τη δυνατότητά τους να ανακάμψουν την δυνατότητά τους να παραμείνουν στην Ευρώπη, να ενδιαφέρονται για την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ευρωπαϊκοί λαοί να νιώθουν αλληλέγγυοι με την Ευρώπη όλων μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντενάνο, συνάδελφε. Η κυρία Γιακοβιέτσκα τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Προεδρία για το έργο το οποίο επετέλεσε. Κυρίως να ευχαριστήσω για το έργο, για την, οδηγίε, τις οδηγίες που είναι οι πιο δυσχερείς, όπως είναι η απόσπαση εργαζομένων. Ήταν το τελευταίο θέμα της ελληνικής προεδρίας αυτό και υπήρχαν πολλές δυσκολίες κυρίως όσον αφορά και το περιβάλλον πριν από την εκλογική αναμέτρηση, αναμέτρηση που κατέστησε δυσχερέστερη την αντιμετώπιση αυτού του χαρτοφυλακίου. Η ελληνική προεδρία στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο λοιπόν κατάφερε να πετύχει ε, κατά 100% την υλοποίηση των προτάσεων. Αυτό είναι σημαντικό. Ο πρόσωπος της προεδρίας ήταν επιτυχέστατος. Η ελληνική προεδρία ήταν εξαιρετική, φαινο, πραγματικά εξαιρετική και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έχουμε απόλυτη υπεποίθηση ότι αυτή η διαφάνεια θα δώσει, θα οδηγήσει στο να επιτευχθούν μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία και αυτό ευχόμαστε να γίνει στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Ζαχμογιέσκα. Τώρα Κώστα έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναγνωρίσω στην ελληνική προεδρία ότι κατάφερα να εργαστεί σε συνθήκες ιδιαίτερων ε, δυσκολιών, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται για μια διαφορετική εποχή της ευρωμεσογειακής πολιτικής ε, λόγω ορισμένων βημάτων που έγιναν. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι μέσω των δικών σας ε, δράσεων ήρθε στο προσκήνιο προσκήνιο ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια πραγματική Ευρώπη δίχως μια μεσογειακή πολιτική και εδώ θα πρέπει να εντάξουμε μια νέα πολιτική πολιτική αλληλεγγύης που να αφορά τη μετανάστευση. Υπάρχει όμως και ένα κεφάλαιο και μια τελευταία ανακοίνωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε ό,τι αφορά θέματα πολιτιστικά. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δίχως άλλο θα υιοθετήσει και η Ιταλική Προεδρία. Αναφέρομαι στο θέμα της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ένα από τους μεγαλύτερους πόρους, ως ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για έναν νέο πολιτιστικό τουρισμό, για μια οικονομία που θα βασίζεται και την πολιτιστική βιωσιμότητα όχι μόνο στην οικονομική και περιοδική. Πιστεύω ότι η προσοχή της ελληνικής προεδρίας που εστιάστηκε σε αυτό το σημείο είναι κάτι που πραγματικά μας ε, ε, απασχόλησε. Πιστεύω ότι υπάρχει μια έλλειψη στη στρατηγική του 2020 και μπορεί να υποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σπυράκη τώρα παρακαλώ. Μικρόφωνο, παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Excuse me, I'm a very ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, η ελληνική προεδρία έδειξε ότι τα κατάφερε, η Ελλάδα έδειξε ότι τα κατάφερε, αλλά τώρα που τα φώτα φεύγουν από εμά, χρειαζόμαστε στήριξη. Χρειαζόμαστε στήριξη γιατί η ελληνική κυβέρνηση, κορμός της οποίας είναι η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που εκπροσωπώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχωρά στις διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις και μία από αυτέ είναι η μερική αποκρατικοποίηση τη ΔΕΗ κόντρα σε παλιού συνδικαλιστέ και την αριστερά. Χρειαζόμαστε όμω στήριξη, χρειαζόμαστε δουλειέ, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε και τα project bonds είναι μια τέτοια ιδέα. Χρειαζόμαστε σταθεροποίηση του οικονομικού τοπίου και η υλοποίηση τη δέσμευση για τη μείωση του ελληνικού χρέου που ελήφθη από του εταίρους μα το Νοέμβριο του 2012 πρέπει να συμβεί άμεσα αφού προηγουμένω ολοκληρωθούν τα stress τεστ των τραπεζών από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα με τους ίδιους όρου και τους ίδιους κανόνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε κυρία Σπυράκη. Ακολουθεί. Ο κύριος Χρυσόγονος, παρακαλώ. Με την ε, πρακτική της η ελληνική προεδρία αναδείχθηκε σε άξιο υπηρέτη της πολιτικής των ευρωπαϊκών ελίτ. ακολουθήσατε την πολιτική της ευπηθούς συμμόρφωσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ίδια που ακολουθείτε σε ελληνικό επίπεδο εκτελώντας τις επιταγές της τρόικας. η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν έφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα για την ευρώπη και αντιθέτως η τραπεζική ένωση την οποία υποτίθεται ότι επιτύχατε στην πραγματικότητα είναι μια τραπεζική διάλυση θα μειώσει την εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες της περιφέρειας ιδίως της ευρωζώνης παρά θα την αυξήσει αλλά και γενικότερα είναι μια πολιτική η οποία μακροπρόθεσμα οδηγεί στη διάλυση της ευρώπης στην κατάρρευση της ευρωπαϊκής ενοποίησης χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική πολιτική μια άλλη ευρώπη μια ευρώπη των λαών και όχι μια ευρώπη των κεφαλαιαγορών την οποία εσείς υπηρετείτε. Ο κύριος για να κλείσει η διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αναδείξω περισσότερο το γεγονός ότι η ελληνική προεδρία πέτυχε αυτά τα σημαντικά που πέτυχε ειδικά στο banking union στην τραπεζική ένωση και στις εργασιακές σχέσεις σε μια περίοδο όπου η χώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και σε μια προεκλογική περίοδο. αυτό αποδεικνύει ότι στάθηκε στεναρά και πειθαρχημένα απέναντι στον λαϊκισμό που επιβεβαιώνει και το εκλογικό αποτέλεσμα ακόμη ότι εάν όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι που θέλουμε να προχωρήσουμε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις για μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα πρέπει όντως να παραμείνουμε σταθεροί απέναντι στον λαϊκισμό. Συγχαρητήρια κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό μα οδηγεί στο να τερματιστεί διαδικασία Catch και δίνω το λόγο στον Επίτροπο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν επισκεφθήκαμε την Ελλάδα στις αρχές της Προεδρίας σας, τονίσατε πόσο σημαντική θα ήταν η Προεδρία αυτή για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα σας την ε, αποκαλέσατε Προεδρία της Επανόδου και αυτή η επάνωδος ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Η χώρα σας επέστρεψε στις οικονομικές αγορές, την ανάπτυξη. Πετύχατε ένα πλεόνασμα μετά από χρόνια και εξ ονόματος της Επιτροπής ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να χρησιμοποιηθεί ακόμα και το τελευταίο τελευταίο λεπτό για να, μπορέσει, να μπορέσουν να περάσουν τα νομοθετήματα που θα έκαναν την Ευρώπη πιο δυνατή. Και δεν συμφωνώ με μερικά από τα σχόλια που άκουσα ότι σήμερα δεν είναι σημαντική η Προεδρία. Η, Προεδρία προεδρεύει σε 9 στα 10 συμβούλια Υπάρχουν πολλές ομάδες εργασίας και ξέρουμε ότι χωρίς την προσωπική δέσμευση και προσπάθεια απλά και μόνο δεν θα μπορέσει να υπάρξει επιτυχής προεδρία. Θα ήθελα συνεπώς να ευχαριστήσω τον Υπουργό σας, τον κύριο Κούρκουλα, τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος κάθεται δίπλα σας και όλους τους εμπειρογνώμονες με τους οποίους συνεργαστήκαμε, γιατί η συλλογική προσπάθεια ήταν αυτή που οδήγησε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πολλοί αναφέρθηκαν στη σημασία της Τραπεζικής Ένωσης, αναφέρθηκαν στην οδηγία για την μετάθεση των, για την απόσπαση των εργαζομένων. Έγινε μια αναφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όλες αυτές είναι πολιτικές όλα τα θέματα που αφορούν εσωτερικές υποθέσεις έχουν συζητηθεί. Όλα αυτά επετέφθησαν χάρη στις προσπάθειες της ομάδας σας, χάρη στην καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επιθυμούσα προσωπικά να ευχαριστήσω στους συναδέλφους σας για την θαυμάσια δουλειά που έγινε προετοιμάζοντας την διάσκεψη κορυφής και συμπληρώνοντας το σημαντικό αυτό χαρτοφυλάκι και που θα παίξει σημαντικό ρόλο για, το, για τις επόμενες εκλογές. Η Προεδρία, αναλάβατε την Προεδρία σε μια κομβική στιγμή για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να πούμε ότι έξι μήνες μετά την ανάληψη της Προεδρίας καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια Ευρώπη πιο ισχυρή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό και να ευχηθώ στην χώρα σας και στους πολίτες αυτής της χώρας ό,τι καλύτερο, αλλά και ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε Σεφτσοβιτς. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ξενόματος ε, του Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς παρακαλώ. Well, I would like to thank, uh... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη για τα θετικά σχόλια που διατύπωσαν για την ελληνική προεδρία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια στρατηγική στρατηγική ασφάλεια, που θα πρέπει να πω ότι συμπεριλαμβάνει και τι θαλάσσιες ζώνες και τον σεβασμό του δίκαιου θαλάσσιου, του δικαίου θαλάσσης. Θα επιθυμούσα επίση να ευχαριστήσω του συναδέλφους που αναφέρθηκαν σε λύσει. Ε, που προτάθηκαν για τις αρχιτεκτονικές ανεπάρκειες της Ευρώπης, εκεί που υπάρχουν. Έχω τη βεβαιότητα, όπως είπε ένα συνάδελφος, δόθηκε πρωτίστως σημασία στην Ελλάδα και όχι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι μερικές ε, ε, απαντήσεις θα έπρεπε να δοθούν. Το 2010, όταν ε, ε, πληγήκαμε από την κρίση. Η Νομισματική Ένωση δεν είχε στη διάθεσή της εργαλεία για την αντιμετωπίση. Η κρίση μας βρήκε απροετοίμαστους. Δεν υπήρχε ESM, SRM, SRM, ε, SRF, τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Και πιστεύω ότι τώρα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αποτρέψουμε μια τέτοια κρίση πριν εμφανιστεί, να την αντιμετωπίσουμε όταν εμφανιστεί. Θα πρέπει να πω ότι αν θα έπρεπε να ξαναγράψουμε και πάλι τον οδικό μας χάρτη μετά από την κρίση, όλοι μας ε, συμφωνούμε ότι θα τον γράφαμε με διαφορετικό τρόπο και εγώ ανήκω σε αυτούς που επέκριναν την πολιτική που υιοθετήθηκε από την αρχή. Αλλά η δική μου θέση ως Πρωθυπουργού της χώρας μετά τον Ιούλιο του 2012 δεν ήταν να επικρίνω τις πολιτικές ή να εμπλακώ σε μια ακαδηματική ακαδημαϊκή συζήτηση για την τέλεια συμφωνία σταθεροποίηση. Το πρόβλημά μου ήταν να διασώσω τη χώρα λαμβάνοντα υπόψη τα λάθη του παρελθόντο και ε, τα διαφορετικά προβλήματα. Αλλάξαμε ό,τι μπορούσε να αλλάξει. Εφαρμόσαμε ό,τι μπορούσε να εφαρμοστεί και καταλήξαμε σε απτά αποτελέσματα. Δεν ήταν εύκολο, ήταν ιδιαίτερα αλγινό και αγαπητοί φίλοι καταφέραμε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει επιτευχθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Διορθώθηκαν τα προβλήματα του ΕΠΕΣ, ε, ε, ε, σταθεροποιήσαμε την καταραίουσα οικονομία, καταλήξαμε σε ένα πρωτογενές πρεώνας ένα χρόνο νωρίτερα βγήκαμε νωρίτερα στις διεθνείς αγορές, πολύ νωρίτερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Και παρόλα τα σοβαρά μέτρα λιτότητας καταφέραμε να ανατρέψουμε την πορεία της ανεργίας, η οποία ακολουθεί μια πτωτική τάση. Βάζουμε τέλος σε μια περίοδο ύφεση εξαιρετούς. Τώρα περνάμε σε μια περίοδο ανάκαμψης και οι προοπτικές υπάρχουν για τη χώρα. Ναι, οι Έλληνες υπέφεραν πάρα πολύ. Ναι, ο λαός στη χώρα μου υποφέρει. Είναι η πρώτη φορά και είναι το πρώτο πράγμα που συνεχίζω να λέω κάθε φορά που συναντώ με ένα ξένο ηγέτη. Τα πράγματα όμως τώρα βελτιώνονται. Σε δύο χρόνια από τότε που αναλάβαμε, σε ε, ανάλαμε πριν από δύο χρόνια. Σε μερικά χρόνια θα είναι απλά και μόνο μία κακή ανάπτυξη. Α πάρουμε το παράδειγμα τη Αργεντινή, μία πλούσια χώρα η οποία πτώχευσε το 2002. 12 χρόνια αργότερα, σήμερα, συνεχίζουν να διανύουν μία περίοδο κρίση και βρίσκονται στο χείλο τη κατάρρευση υποφέρουν πολύ περισσότερο και αυτό είναι κάτι που δεν θα θέλαμε να συμβεί στην Ελλάδα και τα καταφέραμε με την οριμότητα και με τις θυσίες του ελληνικού λαού και με την αποφασιστικότητα που επέδειξε η κυβέρνησή μου. Μερικοί δεν ήθελα να αλλάξει απολύτως τίποτα στην Ελλάδα. Μερικοί καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να βάλουν προσκόμματα στι αλλαγές, στις ιδιωτικοποίησεις, για να τρομοκρατήσουν τους επενδυτές, για να κρατηθούμε στην παγίδα αυτή. Ορισμένοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική κρίση σαν μια πρόφαση για να βγούμε από το ευρώ ή να χρησιμοποιήσουν τα αρχιτεκτονικά ε, προβλήματα της Ευρώπης σαν πρόφαση για να καταρρεύσει όλη η Ευρώπη. Δεν τους αφήσαμε να το κάνουν και πραγματικά είμαστε περήφανοι που δεν τους αφήσαμε γιατί τα πράγματα βελτιώνονται στην Ελλάδα καθώς βγαίνουμε έξω από την ε, σοβαρότερη κρίση που έπληξε την χώρα μας και θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένους ευρωβουλευτές ε, και να τους πω ότι δεν έχω την υποχρέωση να απαντήσω σε ακραίους και δημαγωγούς. Εγώ εξυπηρετώ τα συμφέροντα της χώρας μου. Δεν θα ζητήσω συγγνώμη σε ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, που δημιουργούν διαρκώς προσκόμματα στους επενδυτές, στις ιδιωτικοποιήσεις και πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με την αξιοπρέπεια της χώρας μου, οποιασδήποτε χώρασα, να ζει με δανεικά. Εμείς βάλαμε ένα τέλος σε αυτό και κάνοντας κάτι τέτοιο νομίζω ότι εξυπηρετήσαμε τα συμφέροντα της χώρας μου. Ακούστηκε κάτι πριν από λίγο η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία και οι δημοκρατίες δεν ε, διώκουν, διώκουν τις δράσεις, δεν διώκουν τις πεπιθήσεις. Ε, οι, τα μέλη της ε, χρυσή Αυγής διώκονται για εγκληματικές πράξεις. Λαμβάνουμε σοβαρά τον νόμο και την τάξη. Δίχως τον νόμο, δίχως την τάξη δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Η χρυσή αυγή διώκεται ως εγκληματική οργάνωση λόγω της υποθέμενης εμπλοκής της σε εγκλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Ναζί ήταν η μεγαλύτερη τύρανοι και δεν είναι αποδεκτοί οι θαυμαστές των Ναζί. Θα πρέπει να επαναλάβω ότι οι ηγέτες διώκονται για αυτό που κάνουν και όχι για τα πιστεύω τους. Διώκονται από την δικαιοσύνη και όχι από την κυβέρνηση. Και έτσι θα πρέπει να γίνεται σε κάθε δημοκρατία στον κόσμο. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι που άκουσα για κάποιον που δεν... Ε, δεν γνώριζε καλά τα πράγματα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μία χώρα μέλος μπορεί μονομερός να ε, απορρίψει τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, όπως αποφασίστηκε πριν από δύο μήνες από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και από το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντας. Ένα τελευταίο σημείο, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την κρίση στην Ουκρανία, η ε, Προεδρία, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, υιοθετούν τη διτή προσέγγιση, πολιτική λύση και περισσότερε κυρώσει, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται. Και θα ήθελα να τελειώσω λέγοντα ότι είμαστε έτοιμοι σε στενή συνεργασία με την επερχόμενη Ιταλική Προεδρία για την επόμενη, το επόμενο εξάμεινο, που έχω τη βεβαιότητα ότι θα είναι και πρέπει να είναι επιτυχή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Ολοκληρώθηκε εδώ αυτή η συζήτηση. Διακόπτεται μέχρι τη μία η ώρα η συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου θα έχουμε την εκλογή των κοσμητόρων.